Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικών. Θα ήθελα καταρχάς να σας πενθυμίσω πως πρέπει να εγκριθεί η ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αλλαγές, η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Σημείο 3 έγκριση των πρακτικών για την συνεδρίαση της 6ης Φεβρουαρίου 2017. Ανακοινώσεις του Προέδρου, σημείο 4. Αφορούν την συνεδρίαση των συντονιστών στην στις 21 Μαρτίου. Στη συνεδρίαση αυτή οι συντονιστές αποφάσισαν να συνταχθεί γνωμοδότηση για την έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, που αφορούν την ένταξη των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την καταπολέμηση των ε, δυσάρεστων συναισθημάτων απέναντι στους τσιγκάνους και να αναλάβει τη γνωμοδότηση η ΓΚΟΕ. Μετά, να συνταχθεί γνωμοδότηση στην έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμού για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, προετοιμάζοντας τη θέση του Κοινοβουλίου για το που μετά το 2020. Η... Τη γνωμοδότηση αυτή θα αναλάβει η ομάδα των σοσιαλδημοκρατών. Μετά, να υποβληθεί μια προφορική ερώτηση για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, ιδιαίτερα για την κατάσταση των γυναικών και των παιδιών. Μετά, ε, έκθεση για την ισότητα των φίλων στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αναλάβει την έκθεση το ΕΛΚ. Μετά, Ανάθεση της έκθεσης για τα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης παρενόχλησης, εκφοβισμού και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στο δημόσιο, στους δημόσιους χώρους και την πολιτική ζωή στους σοσιαλδημοκράτες. Μετά η κυρία Μαρία Αρενά να γίνει επικεφαλής της αποστολής της Επιτροπής Γυναικών στην Πολωνία ε, από τις 22 στις 24 Μαΐου. Μετά η επόμενη απόφαση των συντονιστών αφορά τις εξής αποστολές και την προτεραιότητα που θα δοθεί σε αυτές για το δεύτερο μισό του 2017. Οι αποστολές θα γίνουν στη Σουηδία, Τουρκία και Πορτογαλία και θα διοργανωθούν ακροάσεις για τα ακόλουθα. Διακιν... Συνάντηση ε, κοινή επιτροπών για τη βία κατά των γυναικών με έμφαση στη, συνθή... στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Μετά η κατάσταση και τα δικαιώματα των γυναικών με αναπηρία, ευρωπαϊκή στρατηγική κατά τους καρκίνους που πλήττουν γυναίκες και συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό και την εφαρμογή του προγράμματος Δάφνη. Μετά αποφασίσαμε στους συντονιστές να καλέσουμε την κυρία Καταρίνα Μαρσελίνο, ε, Υπουργό Εσωτερικών της Πορτογαλίας, υπεύθυνη για θέματα ηθαγένειας και ισότητας σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις μας. Αυτά λοιπόν ως προς τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές και αυτά ως προς τις ανακοινώσεις που είχα να σας κάνω. Περνάμε στο σημείο 5, η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για τα αποτελέσματα της 61ης Συνόδου Επιτροπή του ΕΕ για τη θέση της γυναίκα, οικονομική χειροφέτηση των γυναικών. Συνσηγήτριε η Κωνσταντ Λεγκρίπ και η Μαρία Αρένα. Αρχίζουμε την ψηφοφορία χωριστή κατά τμήματα. Πρώτο κομμάτι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται τελική ψηφοφορία. Α, δεν χρειάζεται τελική ψηφοφορία, εγκρίθηκε. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Και προτείνω να περάσουμε στο σημείο 6 όπου θα καλωσορίσουμε την κυρία Μύρια Βασιλιάδου, Ευρωπαία Συντονίστρια για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Βασιλιάδου, έτσι ώστε να μας παρουσιάσει την τελευταία έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Έχετε το λόγο κύριε Βασιλιάδου. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ξέρω ότι γίνονται ταυτόχρονα πολλά ενδιαφέροντα ε, στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που στηρίζει το έργο κατά της εμπορίας ανθρώπων. Οι βουλευτέ μας έχουν βοηθήσει, υποστηρίξει και το θέμα παραμένει στην ημερησία διάταξη. Επικαιρών είχαμε δύο ψηφίσματα το 2016 για το εμπόριο ανθρώπων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία παρακολουθούμε μάλιστα εκ του σύνδικης. Γνωρίζετε πολύ καλά πως υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εμπορία. Έχουμε την οδηγία και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την εκρίζωση της ε, εμπορίας προς ανθρώπων που έλξε το τέλος του 2016. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω σήμερα, πολύ συγκεκριμένα, είναι να σας παρουσιάσω δύο από τις τρεις εκθέσεις ε, που δημοσιοποίησε η Κομισιόν το 2016 σε σχέση με την οδηγία. Η πρώτη έκθεση ήταν η πρώτη έκθεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόοδο στον τομέα τη καταπολέμηση εμπορία ανθρώπων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι άλλε δύο εκθέσει έχουν να κάνουν με τη μεταφορά τη οδηγία στο εθνικό δίκαιο και βέβαια έχουμε και την έκθεση των χρηστών. Αυτέ είναι δύο εκθέσει για τι οποίε έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ξεκινήσω σε ένα λεπτό με αυτά. Όμω προ το παρόν να πω κάτι άλλο. Η σημερινή στρατηγική, όπως είπα, έληξε. Είχαμε 40 δράσεις αυτή τη στρατηγική, 38 ήδη έχουν ολοκληρωθεί. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής. Πέρυσι είχαμε πέντε μελέτες μεγάλης κλίμακας που ολοκληρώθηκαν για το φίλ, για τα παιδιά, ε, για μελέτες περιπτώσεων εργασιακής ε, ε, ε, εκμετάλλευσης, χρηματοδότηση, θα σας πω κάποια παραπάνω για το τελευταίο θέμα και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι από τη στιγμή που εγκρίναμε την πρώτη στρατηγική το 2012 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Είχαμε την χρηματοπιστωτική κρίση, τις προκλήσεις με το μεταναστευτικό, απειλές ε, στον τομέα της ασφάλειας, ε, διακρατικά και το πολύπλοκο αυτό φαινόμενο της ε, διακίνησης ανθρώπων. Μεγαλύτερη λοιπόν ε, ευαλωτότητα για τα διακινούμενα άτομα. Αύξηση λοιπόν των θυμάτων από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Το μόντους operandi έχει αλλάξει. Έχουμε αύξηση της διακίνησης για σεξουαλική εκμετάλλευση, πάντα στο πλαίσιο του μεταναστευτικού. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλος κόμβος ε, διακινητών και λατρεμπόρων ε, η Μεσόγειος και επίσης ξέρουμε ότι η διακίνηση ανθρώπων, η εμπορία ανθρώπων δεν έχει να κάνει μόνο με το οργανωμένο έγκλημα, όπως αναφέρεται στη συνθήκη, αλλά στη συνθήκη αναφέρεται η σχέση και με την παρά μετανάστευση. Και βέβαια έχουμε και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ρητός ε, προβλέπει ότι πρόκειται για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σήμερα η εμπορία ανθρώπων και το μετά το 16 πλαίσιο αναφέρονται στην Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, Θεματολόγιο για την Ασφάλεια, στην στρατηγική μας για μια πολιτική ασφάλεια και άμυνα, στο σχέδιο δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο νέο πλαίσιο των δραστηριών της Ένωσης ε, για την ε, ισότητα των δύο φύλων και τη χειραφέση των γυναικών, το 2016 στο 2020. Και στη στις προσπάθειες, ε, τις στρατηγικές για την ισότητα των φύλων. Πολλές λοιπόν αναφορές για τα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά την εμπορία ανθρώπων και τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Τι λέει η Europol. Η Europol στον περασμένο μήνα που έχει εξετάσει τις βασικές απειλές λέει ότι η διακίνηση των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σημαντική απειλή. Δεν θα επεκταθώ στο πώ ε, πραγματεύεται το θέμα αυτό. Η Europol μπορεί να διαβάσετε την έκθεση. Γνωρίζουμε όμως ότι είναι προτεραιότητα και στον κύκλο πολιτικής της Ένωσης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θεωρούν ότι είναι προτεραιότητα το ίδιο και η Europol, το ίδιο και η Κομισιόν. Και σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε. Με βάση λοιπόν τη δική σας έκθεση, την έκθεση του Κοινοβουλίου για την οδηγία του 2011, εγώ θα σας παρουσιάσω τη δική μας έκθεση για την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Αυτό είναι το επόμενο θέμα. Λοιπόν, τι λέει η επόμενη διαφάνεια. Αυτό είναι το πρώτο νομοθέτημα ποινικού δικαίου μετά τη Λισαβόνα. Πρέπει να είμαστε περήφανοι όλοι μας για το πόσο καινοτόμο, συνεκτικό, πλήρε είναι αυτό το νομικό μέσο γιατί έχει να κάνει με όλα τα θέματα, τη δίωξη, τη βοήθεια, την προστασία, την πρόληψη κτλ. Η προθεσμία ε, έχει εκπνεύσει ήδη από τον Απρίλιο, τις 6 Απριλίου 2013. Και τι έχουμε κάνει. Τον Δεκέμβριο του 2016 δημοσιοποίησαμε μια έκθεση. Αφορά αυτή μόνο την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και όχι την υλοποίηση, όχι την εφαρμογή. Και φυσικά και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τι διαδικασίε σε εθνικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί η πλήρη ε, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, η πλήρη υλοποίηση και ή, αν χρειαστεί θα κινήσουμε διαδικασίε επί παραβάση. Και Βέβαια είμαστε στη διάθεση των χώρων για να τις βοηθήσουμε στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Η έκθεση βασίζεται στα εθνικά μέτρα που κοινοποιούν επισήμως τα κράτη-μέρη στην Κομισιόν. Είχαμε τη μελέτη περί ε, μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εκεί βασιστήκαμε. Τα κράτη-μέλη έδωσαν τη γνώμη τους, υπήρξε διαβούλευση. Τι γνωρίζουμε και αυτό νομίζω έχετε ε, να συμφωνήσει με την δική σας έκθεση για τη μεταφορά της οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο. θα επεκταθώ σε κάθε ένα μέτρο ξεχωριστά και τι κάνει η Κομισιόν για να κερδίσω χρόνο. Θέλω να τονίσω όμως αυτά που γνωρίζουμε. Και τι χρειάζεται. Χρειάζεται περισσότερη πρόοδο σε μερικά πράγματα. Πρώτον, στα ειδικά μετά προστασία των παιδιών. Επίκαιρο ε, είναι κάτι που ανακύπτει συνεχώς και το έχουν υπογραμμίσει πολλές φορές και οι βουλευτέ. Επίσης, ό,τι αφορά το τεκμήριο της ε, παιδικής ηλικίας και την αξιολόγηση ε, της ε, παιδικής ηλικίας. Πριν κινήσουμε κάποια ποινική διαδικασία και επειδή θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά στις ποινικέ διαδικασίες, πρέπει να ορίσουμε τη διαχωριστική γραμμή. Από πότε ένας άνθρωπος είναι παιδί κτλ. Και πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στα παιδιά από ό,τι μέχρι τώρα. Θα πρέπει να δούμε επίση το θέμα τη μη τιμωρία ή ε, τη μη εφαρμογή ποινών. Τα θύματα δεν πρέπει να τιμωρούνται για τα εγκλήματα που χρειάστηκε να ε, κάνουν παρά τη θέλησή τους ε, όσο τα εκμεταλλεύονταν. Δεν υπάρχει θέμα συγκατάθεσης αυτών των ανθρώπων, των θυμάτων. Θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στη βοήθεια, στην παροχή υποστήριξη στα θύματα και στα μέλη τη οικογένεια ε, του παιδιού, του θύματο. Τέλο, και εξίσου σημαντικό, η πρόσβαση σε ανεφόρον παροχή βοήθεια. Η Κομισιόν μαζί και με τους φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν πολλά. Θα επανέλθω, αν χρειαστεί. Η αποζημίωση είναι ένα τομέα που πρέπει να προσεχθεί και πολύ περισσότερα πρέπει να γίνουν στον τομέα τη πρόληψη και τη μείωση τη ζήτηση. Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, κατάρτιση των ε, ειδικών αξιωματών κτλ. κτλ. Δεν κάνουμε αρκετά. Δεν πάμε αρκετά μακριά όσο θα έπρεπε. Έχουν κάνει σημαντικέ προσπάθειε τα κράτη-μέλη για να έρθουν σε συμπεράσματα και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το κατανοήσουμε. Αλλά πρέπει να γίνουν και πολλά ακόμη. Πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την οδηγία για να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση. Επίσης, ε, εφόσον χρειαστεί, θα ε, κινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση, όπως είπα, και επίσης θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης κατευθυντηρίων γραμμών για την ε, πρακτική εφαρμογή της οδηγίας για συγκεκριμένε διατάξει. Ε, βεσικά είναι διαθέσιμη εκθεσή μα, κοινοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο και υπάρχει μια παράγραφο τη οδηγία που είναι άκρω πολύπλοκη. Το άρθρο 23.1 Transposition Measures και το 23.2 of existing national law establishing as a criminal offence the use of services which are the objects of exploitation of trafficking human beings. Πρέπει να το πω τον τίτλο όλο, για να δείτε στα αγγλικά περί τίνος πρόκειται. Έχουμε λοιπόν αυτό το άρθρο, αλλά έχουμε και το άρθρο 19 τρέποστα από τα κράτη-μέλη, τουλάχιστον να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψη μέτρων ε, για να θεωρηθεί αξιόπινη πράξη κτλ. Δημοσιοποίησαμε λοιπόν αυτή την έκθεση το 2016. Θα έλθω σε περισσότερε λεπτομέρειε. Πρώτα απ' όλα, τι κάναμε. Έχουμε την περιγραφή τη Ριστάμενη εθνική νομοθεσία για την ποινικοποίηση τη ε, χρήση υπηρεσιών και αξιολογούμε τον αντίκτυπο των μέτρων. Τι δεν κάναμε όμω με την έκθεση. Δεν εξετάσαμε άλλα μη νομοθετικά μέτρα, ούτε νομοθετικά μέτρα που δεν άπτονται τη ποινικοποίηση τη χρήση των υπηρεσιών. Αυτά κάναμε και αυτά δεν κάναμε. Στείλαμε το ετοιματόλευε στα κράτη-μέλη το Μάιο του 2016. Λάβαμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες από την κοινωνία των πολιτών, την οποία θέλω και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ μέσω της πλατφόρμας 100 ΜΚΟ και βέβαια η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ε, εμπορία ανθρώπων έδωσε και αυτή τη δική της, το δικό της input. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, διάφορες πρακτικές. Και τα κράτη-μέλη λένε είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος. Το 2013 έληξε η προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, έχουν ληφθεί τα μέτρα αυτά στο μεταξύ, αλλά λένε τα κράτη-μέλη δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμη σωστά την κατάσταση. Και περιορίζεται το πεδίο μόνο σε αυτούς που άμεσα κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών των θυμάτων. Δέκα μόνο τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν θεσπίσει τη χρήση πληροφοριών ε, υπηρεσιών συγγνώμη, ως ποινικό αδίκημα. Βλέπετε ποια είναι αυτά. 14 δεν έχουν ε, θεωρήσει ποινικό αδίκημα τη χρήση υπηρεσιών. Τρία κράτη-μέλη, μόνο τρία, για μόνο μία μορφή έχουν ε, πει ότι είναι ποινικό αδίκημα. Αλλά ακόμη και αν δεν υπάρχει διάταξη που να ποινικοποιεί τους χρήστες. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι συχνά τα θύματα έχουν επανειλημμένως υποστεί βιασμό, σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση, περιορισμό ελευθερίας, ε, περιορισμό της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης και της σωματικής του Σταματώ εδώ, αλλά θα πω λίγο παραπάνω. Είναι πάρα πολύ κερδοφόρο το αδίκημα αυτό της διακίνησης ανθρώπων, από τα πιο κερδοφόρο. 29,4 δισεκατομμύρια λέει η Ευρωπόλη είναι το ετήσιο κέρδος μόνο για τους διακινητές. Είναι μηχανή που κόβει πολύ χρήμα. Και για το νομικό κλάδο που ασχολείται με παράνομες αστέτες, αλλά και για παράνομους κλάδους που ασχολούνται με νόμιες δραστηριότητε. Υπάρχει κέρδος και υπάρχει ζήτηση για όλες αυτές τις μορφές εκμετάλλευσης. Είπα επίσης ότι η μετανάστευση έχει δημιουργήσει μια τάση λίγο πολύ σε ό,τι αφορά τι μεταναστευτικέ ζωέ και το πώ αυτέ σχετίζονται με τη διακίνηση ανθρώπων. Η Διεθνής Οργάνωση Μετανα... Ο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση λέει ότι μόνο για το 2016 είχαμε 11.000 γυναίκε και κορίτσια που αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν από την Ιγυρία μέσω της Λιβύης και να πάνε στην Ιταλία όπου και έγιναν ένα ανθρώπινο εμπόρευμα που διακινείται ανά την Ευρώπη. Δεν είμαι και πολύ καλή στα μαθηματικά, αλλά αν κάνω λίγα σπράξεις εδώ αριθματικές θα πούμε 11.000 μέσα σε ένα χρόνο. Έχουν εντοπιστεί. Τι έγινε τα προηγούμενα τρία χρόνια ή τα τελευταία τρία χρόνια και ποιοι είναι πραγματικοί αριθμοί. Τουλάχιστον 10 χρήσει το τη μέρα. Θα μπορούσε να πει κανεί. Α πούμε 300 μέρε το χρόνο. Αν το πολλαπλασιάσουμε αυτό με 11.000 γυναίκε και παιδιά, τι μα δίνει αυτό. Α πούμε δε ότι είναι και φτηνό. 30-40 ευρώ που δεν είναι. Τη φορά. Πού πάνε αυτά τα χρήματα, πού είναι. Η μεγάλη προτεραιότητα για την Κομισιό είναι να ακολουθήσει το δρόμο του χρήματος για να βρει πού πάει στην αλυσίδα της διακίνησης. Τα χρήματα αυτά δεν είναι αυτά τα 30-40 ευρώ μιας ανταλλαγής μεταξύ ενός χρήστη ε, και ενό θύματος. Αλλά υπάρχει διακίνηση, κάποιος μεταφέρει το θύμα, υπάρχουν λαθρέμποροι, σωματέμποροι καλύτερα κάποιοι άλλοι που δευκολύνουν, κάποιοι μεσάζοντες, ε, κάποιοι που κλείνουν τα μάτια σε ό,τι αφορά, χάρη, τη φιλοξενία, το που φιλοξενούν. Και πολλοί άλλοι που βλέπουν τον, ε, μπροστά του στον δρόμο να γίνονται κάποια πράγματα και κλείνουν και αυτά τα μάτια. Άρα θέλουμε να δούμε πού πάει το χρήμα και ποιοι είναι αυτοί που αγοράζουν αυτούς τους ανθρώπους. Σίγουρα είναι σαφείς περιπτώσεις διακίνησης, εμπορίας και άμα βλέπουμε μια νεαρή γυναίκα στον δρόμο, εύκολα καταλαβαίνουμε τι τη συμβαίνει. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Και πρέπει να πω το εξή. Εάν δεν ποινικοποιήσουμε αυτού που εν γνώση τους χρησιμοποιούν τα θύματα, τι κοινωνία δημιουργούμε. Δημιουργούμε μια κουλτούρα ατιμορρησίας στις κοινωνίες μας. Λέμε ότι δεν έγινε και τίποτα. Το πιο απλό μπορεί να πει κανεί είναι ότι μα είναι τόσο δύσκολο να αποδειχθεί. Και υπάρχουν ε, και εισαγγελίε πολύ δεκεκριμένοι, που του σέβομαι και που λένε δώστε μου, πείτε μου ένα έγκλημα που είναι εύκολο να αποδειχθεί. Νομίζω ότι όλε οι μορφές οργανωμένου, σοβαρού οργανωμένου εγκλήματο είναι δύσκολο να αποδειχθούν. Αυτό όμω αποτελεί δικαιολογία για να πούμε ότι δεν θα νομοθετήσουμε. Σχετικά. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να μα απασχολήσει πολύ περισσότερο. Ακόμη και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει μια σύμβαση ε, για τη δράση, για την καταπολέμηση της διακίνησης και λέει ότι η δυσκολία ε, να βρεθούν αποδεκτικά στοιχεία δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να θεωρήσουμε τέτοια συμπεριφορά στο ποινικό αδίκημα. Ολοκληρώνοντας λοιπόν έχουμε διάφορα ε, τοπία, διαφορετικά μοτίβα. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα τιμωρησίας, ούτε από κανονιστικής πλευράς αλλά και γιατί πρέπει να αποτρέψουμε αυτά τα εγκλήματα και επίσης πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ε, λογοδοσία. Θα είναι υπόλογοι οι δράστες και οι χρήστες. Και όταν μιλάμε για τους χρήστες, δεν είναι απλά το ότι ορίστε εγώ αγόρασα αυτό το μπουκάλι που το έφτιαξε ο τάδε που ήταν θύμα κτλ. Όχι. Έχουμε τους μεσολαβητέ του ε, στην αγορά εργασία, έχουμε την αλυσίδα εφοδιασμού, έχουμε τους αξιωτικού πράκτορες, έχουμε τις μεταφορικές εταιρείε. Πρέπει να ξέρουμε ότι για τη διακίνηση έχουμε μια λυσίδα ε, νόμιμων ε, επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αυτά τα κυκλώματα και αποκομίζουν κέρδο. Άρα θα πρέπει όταν νομοθετήσουμε να ξέρουμε γιατί νομοθετούμε, για ποιο νομοθετούμε και κατά ποιού νομοθετούμε. Θέλουμε να μειώσουμε την ζήτηση ε, και να αποτρέψουμε τη δικίνηση. Τι κάνουμε για αυτούς τους τόκους. Βλέπουμε τις πιθανές επιλογές για το μέλλον. και οι δυνατόν όπως αποφάσισαν νομοθέτες μπορεί και να προτείνουμε συγκεκριμένες νομοθετικές ε, προτάσεις. Πριν κλείσω, να μιλήσω για κάτι που το θέτεται πολλές φορές με τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις ε, και σε κάτι ακροάσεις για το χρήμα που το ανέφερα και εγώ, όχι μόνο για τους εκκινητές, αλλά και για τα χρήματα των φορολογουμένων. για να έχουμε μια σωστή πολιτική κατά της διακίνησης. Τι κάναμε έχουμε την ε, αναθεώρηση της ε, συνολικής προσέγγισης. Κάναμε μια χαρτογράφηση της διανομής των έργων από το 2013 μέχρι σήμερα. Τι κάναμε και τι ε, ανακαλύψαμε. Είδαμε όλες τις υπηρεσίες κομισιών τα τελευταία 12 χρόνια τι έχουμε χρηματοδοτήσει. Είδαμε ποιοι ήταν οι δικαιούχοι. Τι ήταν το επίπεδο χρηματοδότηση, ποιο ήταν το output, ποιε ήταν οι συστάσει για λήψη μέτρων πολιτικών και άλλα και μετά είδαμε. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη συνεκτικότητα, να δαπάνονται σωστά τα χρήματα, να έχουν έναν σωστό αντίκτυπο. Βρήκαμε 321 έργα, 160 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν μιλώ για την κρίση μεταναστευτική, γιατί εκεί είναι τουλάχιστον διπλάσια τα ποσά για τα οποία μιλάμε. Πριν τη μεταναστευτική κρίση λοιπόν και από την περίοδο 2004 και μετά, είχαμε 160 περίπου, 160 εκατομμύρια ευρώ. 57% των σχεδίων ε, είχαν ε, ΜΚΟ ε, ως επικεφαλής, το 70% ήταν πριν στρατική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλη αυτή την περίοδο πάνω από το μισό των ποσών το διαχειρίζονταν ΜΚΟ και αυτό θεωρούμε πάρα πολύ καλό. Βλέπουμε επίσης πολλά χρήματα να πηγαίνουν σε διεθνείς οργανισμούς και μιλάμε και για τα πιο σημαντικά έργα. 40 ε, βασικοί ε, επιχορηγούμενοι ε, είχαν πάρει πολλαπλά έργα. Βλέπετε ποιοι είναι, με τα κόκκινα. Κάτι ενδιαφέρον είναι ότι 8 από τους μεγάλους αυτούς επιδοτούμενους πήραν επαναλημμένα χρηματοσία, 5 και παραπάνω έργα. Τέσσερι ήταν μικιό on the road and Το περισσότερα ποσά σε ποσοστά πήγαν στην Αυστρία, αλλά συμπεριλαμβάνονταν και διεθνεί οργανώσει. Μετά Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και 100 Θέλω να κλείσω με κάτι που μα άνοιξε τα μάτια. Και η μελέτη αυτή ήταν πολύ χρήσιμη στα αποτελέσματά της. 56% ε, της χρηματοδότησης πήγε σε διάφορες μορφές, αλλά μη διευκρινισμένες. Πάντως, για την εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού, είδαμε τα περισσότερα να χρειάζονται για τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Η διακίνηση σε σχέση με τη σεξουαλική εκμετάλλευση πήρε τη λιγότερη χρηματοδότηση, αλλά και τα ποσά αναπρόγραμμα. Και είναι πολύ ενισχυτικό. Διότι με όλες τις τάσεις, με όλα τα στοιχεία που είχαμε συγκεντρώσει από την Europol, την UNHCC και ούτω καθεξής, διαπιστώσαμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διακίνηση σε σχέση με τη σεξουαλική εκμετάλλευση, με το 1 τρίτο των ε, θυμάτων. Ε, του αφορά αυτό. Και μόνο 20% της ε, ε, χρηματοδότησης πήγε για γυναίκες, παιδιά και την ε, εμπορία γυναικών. Πρέπει να αποκομίσουμε μαθήματα από αυτό. Να σκεφτούμε καλά το μελλοντικό πολιτικό πλαίσιο που μας ενδιαφέρει. Λιγότερο από το 20% όλων των προγραμμάτων επικεντρώνονται στο φύλλο. Και νομίζω ότι το λέω στη σωστή επιτροπή αυτό. Για μας, ένα λεπτάκι χρειάζομαι για μας αυτό ήταν μια προσπάθεια να διαπιστώσουμε τη λογοδοσία. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Λογοδοσία όχι μόνο για όσα κάνουμε, αλλά και για όσα λέμε. Θα ήθελα να κλείσω με αυτό, τα πόσα λέμε. Ε, παρατηρούμε ότι όλο ένα και περισσότερο έχουμε ένα καλάθι. Και επειδή είναι πολύ τώρα, μιλάμε για κρίσεις όλα τα επίπεδα, οπότε τι κάνουμε στο καλάθι βάζουμε πολλούς διαφορετικούς όρους. Διακίνηση, σκλαβιά, δουλεία, ε, ξεναγκιστική εργασία, καταναγκαστική μάλλον εργασία, λαθρεμπόριο, όλα στο ίδιο καλάθι. Μερικοί όροι από αυτούς δεν είναι καν ε, νομικοί ορισμοί, είναι επικοινωνιακά εργαλεία. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα θύματα, και αν θέλουμε να διώξουμε του ε, δράστε ή του αυτούργου, πρέπει να έχουμε νόμου και να είναι σαφεί και ορισμοί. Και δεν μπορούμε αυθερέτως να χρησιμοποιούμε λέξεις όπως ε, σύγχρονη σκλαβιά και δουλεία, καταναγκαστική εργασία, λαθρεμπόριο και διακίνηση και εμπορία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχει σημασία διότι αν δεν εντοπίσουμε το πρόβλημα δεν μπορούμε να βρούμε και λύσεις. Και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό ω πολιτικοί ηθήνοντε που είστε. Ε, και θα ήθελα λοιπόν κλείνοντα να κάνω το ίδιο, να πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Διαβάζοντα την εφημερίδα, βλέπω ότι υπάρχει ένα άρθρο για την διακίνηση και λέει όλο καταναγκαστική εργασία, ε, λαθρεμπόριο. Ε, ο τίτλο λέει εμπορία ανθρώπων και δεν έχει καμία σχέση με το θέμα. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μιλούμε ορθώ και να χρησιμοποιούμε του σωστού νομικού ορισμού. Αυτό που θα κάνουμε τώρα λοιπόν είναι να καταρτήσουμε ένα πολιτικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2016, όπως προέκυψε από τι συζητήσεις μας, να εξετάσουμε τι μορφή θα πάρει αυτό, να το δούμε προσεκτικά στην Επιτροπή, γιατί το συζητήσαμε διεξοδικά με του εξωτερικούς ενδιαφερομένου. Σας ευχαριστώ για τα ψηφίσματά σας, διότι θεωρώ ότι είναι ένα απόσπαστο τμήμα των όσων πρέπει να μας απασχολήσουν όπως προχωρούμε και ελπίζω να, με, να, είστε μαζί μου όταν ε, κάνουμε την προσπάθεια για να εντοπίσουμε τα θύματα της διακίνησης ε, που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε από πέρσι. Τα παιδιά των 8 ετών και να αναρωτηθείτε ποια είναι τα παιδιά, ε, ποια είναι τα θύματα, συγγνώμη. Ε, μας ενδιαφέρει ποια είναι τα θύματα αλλά και ποιοι είναι αυτοί που ωφελούνται, που αποκομίζουν κέρδος από την ε, διακίνηση. Τι θα κάνουμε για να εντοπίσουμε τους εγκληματίες, τους δράστες, τους αυτούργους, το χρήμα που προκύπτει ποιοι είναι αυτοί που είναι αντικείμενο εμπορία, αγόρια και κορίτσια, αλλά όχι μόνο, και πώς το κέρδος αυτό, το οικονομικό, ε, τελικά αναζω, την ε, ζήτηση. Αυτά θα μας απασχολήσουν και θα απασχολήσουν και την Επιτροπή σας τα ερχόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Βασιλιάδου. Και τώρα να ξεκινήσει η συζήτηση με τους συναδέλφους. Η κυρία Ρενά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Είναι εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Ακούτε, ακούτε τη διερμηνία. Ακούγεται η διερμηνία στα ελληνικά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, η οποία ήταν πολύ επικοδομητική. Και συμφωνώ μαζί σα, Δεν λέμε τα πράγματα με το σωστό όνομα, το σωστό όρο. Δεν έχετε διερμηνία. Με ακούτε. Με ακούτε. Με ακούτε εντάξει. Έχετε διερμηνία. Με ακούτε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ήθελα λοιπόν να σας θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το φαινόμενο της μετανάστευσης. Όταν μιλάμε για τη μετανάστευση, συναντούμε όλες τις μορφές τις οποίες αναφέρατε. Που λειτουργούν σωρευτικά. Έχουμε δηλαδή από τη μια το λαθρεμπόριο, Έχουμε τους διακινητές, έχουμε την ίδια την εμπορία, την εμπορία ανθρώπων, Έχουμε το φαινόμενο της εκμετάλλευσης και της καταναγκαστικής εργασίας. Έχουμε το φαινόμενο της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Έχουμε το θέμα του ευάλωτου κοινού, των ευάλωτων ομάδων δηλαδή, τα παιδιά, οι ασυνόδευτοι ενήλικοι και οι γυναίκες. Άρα στα πλαίσια της μετανάστευσης υπάρχουν περίπλοκα υποφαινόμενα που συνδυάζονται και έχουν να κάνουν με την ε, διακίνηση των ανθρώπων. Ε, Ήθελα να μου πείτε κατά πόσον η οδηγία για την εμπορία των ανθρώπων ε, μπορεί να εφαρμοστεί ακριβώ το φαινόμενο τη μετανάστευση. Τι μπορούμε να κάνουμε για να είναι πιο δραστική και αποτελεσματική. Και τι άποψη έχετε για τι συμφωνίε που έχουν συνάψει τα κράτη-μέλη με χώρε εξωτερικέ τη Ένωση. Δηλαδή η συμφωνία με την Τουρκία, αλλά και η Ιταλία ετοιμάζεται να συνάψει συμφωνία με τη Λιβύη χώρα η οποία δεν σέβεται καθόλου τη σύμβαση της Γενέβη, Και ούτε υπόκεινται στην οδηγία μας προφανώς, αλλά ούτε καν στις συμβάσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ισχύουν διεθνώ. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να απαιτήσουμε από τα κράτη-μέλη που ετοιμάζονται να συνάψουν συμφωνίες με εξωτερικές χώρες να ε, ζητούν εγγύησεις. Εγγύησεις ώστε αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατάχρηση, για να το πω έτσι, την ε, εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών που εμπλέκονται στο φαινόμενο της μετανάστευσης να πάψουν. Ε, υπάρχει εξωτερήκευση, εξωτερική ανάθεση ουσιαστικά τη αντιμετώπιση του φαινομένου και τη εκμετάλλευση των ευάλωτων ομάδων. Στο πρώτο σκέλο αυτό. Στο δεύτερο, προσφάτως στις εφημερίδες, ήδη το 2015 δηλαδή, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο για τις γυναίκες γεωργούς στη Σικελία. Τις γυναίκες που απασχολούνται στη γεωργία στη Σικελία που είναι από τη Ρουμανία. Είναι πολύ κινητικές εντός της Ευρώπης, αλλά είναι θύματα και της καταναγκαστικής εργασίας με συμβάσεις που είναι συμβάσει οι οποίε καθόλου δεν σέβονται του όρου των συμβάσεων τη Ευρώπη, αλλά και με την σεξουαλική εκμετάλλευση. Δηλαδή, ισχύει μια μορφή σεξουαλικής ε, σκλαβιάς όπως είχε τον 19ο ε, αιώνα. Η οδηγία για την ε, εμπορία των ανθρώπων λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόζεται. Πώ πώς μπορείτε να κάνετε την αξιολόγηση της υλοποίησης της οδηγίας που είναι υποχρεωτική από το 2013 και πώς μπορεί να υπάρξει ε, προσφυγή των ανθρώπων αυτών για αυτές τις ε, κακοποιήσεις και μορφές εκμετάλλευση στο πλαίσιο της ε, ισχύουσας υποτίθεται οδηγίας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκέορκ, κυρία Μπιόρκ, συγγνώμη, και αν μπορείτε να είστε σύντομοι, διότι έχουμε και άλλα σημεία στην μέση διάταξη. Ευχαριστώ, δεν θα με ακρηγορήσω. Το πήρα το μήνυμα. Ήθελα να ευχαριστήσω τη συντονίστρια για την εμπορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι νομίζω ότι ήρθατε με πολύ σαφή μηνύματα, με καταγραφή στοιχείων, με συλλογή δεδομένα από όλε τι εκθέσει. Ελπίζω πραγματικά η Επιτροπή συνολικά, εσείς και ο Επιτροπός μας, ο κ. Αβραμόπουλος, να προχωρήσετε σε στενή συνεργασία με την κυρία Γιούροβα, που είναι υπεύθυνη για την ισότητα των φύλων, ότι θα προχωρήσετε και θα πάρετε τα απαραίτητα μέτρα για την κατάρτιση μιας ευρωπαϊκής Ε, Πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερω τι προσπάθειέ σα. Χρειαζόμαστε πρόοδο και στα δικαιώματα των παιδιών, στην ε, προστασία, στην ε, ε, απομονή δικαιοσύνη για τα θύματα, την αποζημίωσή του, την πρόληψη και την προστασία των υστέρων και επίση καταγράφω με κάποια ανησυχία την ότι τα προγράμματα είναι κάπως ε, χαλαρά ε, και όχι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της εμπορίας. Θα θέλαμε όντως αποτελέσματα, χειροπιαστά αποτελέσματα. Εκεί προσπαθούμε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και ελπίζω μελλοντική στρατηγική να, να επικεντρώνεται περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών και την προστασία των θυμάτων. Και την πρόληψη. Δεν λέω ότι η δίωξη δεν είναι σημαντικό σκέλος, όμως είναι πολύ οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία και δεν έχουμε δώσει ακόμα αρκετή έμφαση στην ε, προστασία και την πρόληψη. Και για όσα είπε η Μαριά για την ε, μετανάστευση, είναι προφανές ότι η εμπορία γίνεται εκεί. Εκεί τιμωρούνται διπλά τα θύματα. Και για την ε, επικείμενη συμφωνία της Λιβύης με την Ιταλία. Έχουμε διαμαρτυρηθεί γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ σαφεί. Και να βεβαιωθούμε ότι η μελλοντική στρατηγική έχει περισσότερη ουσία για το τέρμα τη ατιμορρησία. Ακόμα και ο όρο χρήστη είναι κακοποίηση, είναι εκμετάλλευση. Δεν μπορεί κανεί να λέει χρήστη. Τι συντηρητική κοινωνία είναι αυτή. Εάν οι άντρε μπορούν να κακοποιούν τι γυναίκε, χωρί να προβλέπεται καν μια τιμωρία, επειδή απλώ υπήρξαν θύματα εμπορία. Και δεν μιλάμε καν για του αρχικού αυτούργου και δράστε. Το ένα πράγμα φέρνει το άλλο δηλαδή και πρέπει το κάθε βήμα να μα οδηγεί στο επόμενο. Οπότε ναι, πρέπει να πάψει η ατιμορρησία των δραστών. Ευχαριστούμε κυρία Νόιφλη. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση προς την εισηγήτρια. Μας ε, αναφέρατε πριν μια διαδικασία παραβάση κατά κάποιων κρατών μελών, μια διαδικασία που θα εφαρμοστεί που εφαρμόζεται όταν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν αρκετά. Εγώ θα ήθελα να μάθω περισσότερα για την κατάσταση στη Γερμανία. Στη Γερμανία, και λυπάμαι που το λέω, υπάρχει ένας πολύ φιλελεύθερος νόμος περιπορνίας και η νομοθεσία αυτή ως αποτέλεσμα, πώς να το πω, έχει δημιουργήσει στη Γερμανία μία ατμόσφαιρα που θεωρεί την πορνεία ένα επάγγελμα όπως όλα τα άλλα. Ε, σίγουρα υπάρχουν εγκλήματα, αδικήματα τα οποία διώκονται, όμως η γενικότερη ατμόσφαιρα που επικρατεί στη χώρα είναι ότι εντάξει μια δουλειά είναι και αυτή. Όσο πιο φιλελεύθερη είναι η νομοθεσία περί πορμηνίας, τόσο πιο έντονη είναι η δράση διάφορων ε, εγκληματικών ε, συμμοριών και τόσο μεγαλύτερη εμπορία ανθρώπων. Ε, θα ήθελα λοιπόν εγώ να ρωτήσω, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ε, το οποίο μπορείτε να κάνετε εσείς κατά της ε, Γερμανίας, να στείλετε κάποια επιστολή, να χρησιμοποιήσετε κάποια διάταξη του νόμου έτσι ώστε να ε, αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Διότι η νομοθεσία αυτή έχει σίγουρα κάποια προβλήματα. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να μάθω τι έχετε να πείτε, διότι σίγουρα η πορνεία δεν μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται ένα επάγγελμα όπως όλα τα άλλα. Έχει κινδύνους που πρέπει να αναφερθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάνιμπολ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Είναι πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τάσετε υπέρ του βόρειου μοντέλου, δηλαδή εκείνος ε, που χρησιμοποιεί, που αγοράζει σεξουαλικές υπηρεσίες, ε, να είναι αυτός που θα διώκεται, να είναι ο ένοχος. Είναι πολύ καλό λοιπόν αυτό το μοντέλο και θεωρώ πως ε, δύο πράγματα χρειάζεται να κάνουμε. Τα έχω αναφέρει και πριν. Έχω αναφερθεί στην επιβολή του νόμου και γνωρίζω πως ε, και εσείς έχετε επαφές με αρχές επιβολής του νόμου. Ήθελα λοιπόν να πω πως καταρχάς ναι, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να διώκουν τους ε, εμπόρους ανθρώπων. Ε, και γνωρίζω πως ανεξάρτητα με τους νόμους περιπονίας η εμπορία ανθρώπων είναι ποινικό δίκημα σε όλα τα κράτη-μέλη. Τι γίνεται λοιπόν εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί, διότι δεν θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο τις εγκληματικές συμμορίες, ούτε να ακολουθήσουμε τον δρόμο του χρήματος, αν δεν ε, ασχοληθούμε με τα προηγούμενα στάδια. Τότε θα είναι αργά. Γι' αυτό ελπίζω να είμαστε σε θέση να ακολουθήσουμε, να εφαρμόσουμε το βόρειο μοντέλο, να το ψηφίσουμε στο Κοινοβούλιο, μια και είναι στην ουσία η πολιτική την οποία πρεσβεύουμε. Διαφορετικά δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθούν τα κρούσματα εμπορίας. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσετε όλο αυτό. Νομίζω πως ε, η δουλειά σας είναι εξαιρετική και καλά κάνετε που μας παροτρύνετε να μην επαναπαυόμαστε, να συνεχίσουμε να συζητάμε το, μένα, ε, το θέμα. Το 3% της ε, χρηματοδότησης, μας είπατε, ε, μόνο πηγαίνει στα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Και η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι ε, ως επιτοπλίστων αυτό που συμβαίνει στα θύματα εμπορίας. Και μάλιστα τώρα με την κατάσταση που επικρατεί με τους μετανάστες και όσους ε, περνάνε τα σύνορα, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Θα ήθελα λοιπόν να το σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλατε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Έχετε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Το πρώτο μήνυμα που θέλω να δώσω καταρχάς είναι ότι τα δύο τρίτα των ε, θυμάτων εμπορίας σύμφωνα με τις τάσεις, με τη γύρω στα την Ευρωπόλ, συνεχίζουν ε, να παραμένουν υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε αν θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα. Μιλάμε δηλαδή για το 80% των θυμάτων που είναι γυναικόπαιδα και ε, οι περισσότεροι από αυτούς δεν, ε, είναι, δεν, ε, μετανάστες, ή πρόσφυγες. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε απόλυτα ενήμεροι για την διάσταση του προβλήματος, έτσι ώστε να μην υπάρχει ατιμορρησία, να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αντιμετωπίσουμε το ίδιο το πρόβλημα. τώρα, σε τη φορά την οδηγία, αφήστε με να πω το εξής. Είναι ένα πολύ καλό μέσο, είναι αρκετά περιεκτική και δεν είναι το πρόβλημα η ίδια οδηγία. Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή της. Η οδηγία παρέχει βοήθεια στα θύματα. Τα θύματα έχουν δικαιώματα. Εμείς αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι να ε, ταυτοποιήσουμε τα θύματα, να εντοπιστούν τα θύματα και να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Και ε, μεταξύ άλλων ο νόμος λέει ότι όλοι οι υπάλληλοι που θα είναι στην πρώτη γραμμή πρέπει να είναι παρκώς καταρτισμένοι για να μπορούν να εντοπίσουν ποιο είναι το θύμα. Είναι όμως καταρτισμένοι. Δεν νομίζω. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τα απαραίτητα μέσα στη διάθεσή μας για να καταρτιστούν οι υπάλληλοι που θα εντοπίζουν αυτά τα θύματα για να μπορούν να τα εντοπίζουν. Και αυτό που χρειάζεται είναι λύση η οποία θα είναι βιώσιμη. Για παράδειγμα, η εξωτερική διάσταση. Εδώ τα κράτη-μέλη ζητείται να κάνουν εκτιμήσεις και εξολογήσεις κινδύνου. Η οδηγία επίσης σέβεται την αρχή της μη επαναπροώθησης. Πρέπει να δούμε εφαρμόζεται στην πράξη. Αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε. Και έχω επίγνωση της κατάστασης στην Ιταλία με τις γυναίκες από τη Ρουμανία και πρέπει να ε, παραδεχτούμε ότι έχουν πέσει θύματα όχι μόνο καταναγκαστικής εργασίας αλλά και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κάτι που περιπλέκει την κατάσταση. Οι διατάξεις υπάρχουν στην οδηγία. Υπάρχει κοινωνία των πολιτών η οποία ε, παρέχει βοήθεια στήριξη, υπάρχει μια ε, ρυθμιστική αρχή, εθνική ρυθμιστική αρχή που συντονίζει τις δράσεις. Η Ιταλία επίσης στην νομοθεσία της έχει πολύ καλές διατάξεις σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των θυμάτων. Το θέμα όμως είναι πώς εφαρμόζεται, κατά πόσο εφαρμόζεται και κατά πόσο είναι αποτελεσματικά τα εθνικά συστήματα ταυτοποίηση των θυμάτων. Χρειάζεται λοιπόν βοήθεια στα κράτη-μέλη και η Ιταλία είναι από τους ε, αποδέκτες βοήθειας αλλά και να γίνουν περισσότερα σε επίπεδο εφαρμογή. Και ας είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με το τι θέλουμε. Υπάρχουν γυναίκες που είναι θύματα εμπορίας ε, καταναγκαστικής εργασίας, υπάρχουν γυναίκες που είναι θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση ε, και όταν είναι θύματα εμπορίας για καταναγκαστική εργασία ποιο είναι το πρόβλημα, ε, οι αμοιβέ, το ωράριο, τι. Επίσης, πρέπει να γίνει μια επανεξέταση του κοινού συστήματος ασύλου, σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο για το άσυλο. Μετά υπάρχει η οδηγία για τις εγκαταστάσεις και τις συνθήκες υποδοχής. Εδώ οι γυναίκες θεωρούνται... Ε, πως δικαιούνται ε, ιδιαίτερες ε, συνθήκες και μετά αναγνωρίζονται οι γυναίκες ως ομάδα ε, που έχει δικές ανάγκες. Μετά, χρειάζεται κατάρτιση για την εμπορία ανθρώπων. Υπάρχουν οι διατάξεις πρώτον για να ε, υπάρχει επαρκής κατάρτιση στους υπαλλήλους που θα αναγνωρίζουν τα θύματα, που θα διεξάγουν μετά τις ε, συνεντεύξεις και που θα βοηθούν τα θύματα σε μια διεθνή ποινική διαδικασία αποζημίωσης. Μετά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν τα μέσα στη διάθεσή μας. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ο έλεγχος της ε, εφαρμογής της νομοθεσίας. Και αυτό αφορά όλους τους φορείς, δυστυχώς. Αυτό έχω να πω. Υπάρχουν ελλείψεις παντού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δίωξη που αναφέρθηκαν νομίζω δεύτερη και τέταρτη μιλήτρια, θα συμφωνήσω. Είναι η κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η δίωξη και η πρόληψη. Νομίζω πως αυτά πάνε χέρι με χέρι, διότι βλέπουμε ότι το χρήμα σχετίζεται άμοσα με τη ζήτηση, η ζήτηση σχετίζεται μέσα με το χρήμα. Σίγουρα χρειάζεται προσοχή και σαφήνεια ε, ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα αναφερόμαστε σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τους άλλους. Δεν πρέπει να τους ε, αναφέρουμε ως πελάτες. Ο πελάτης είναι κάποιος που αγοράζει ένα προϊόν. Το, ένα νεφρό δεν είναι προϊόν που αγοράζεις. Και πρέπει λοιπόν να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα σε πελάτες, σε χρήστες και σε αυτούς που κάνουν κατάχρηση αυτών των όρων. Αυτό που πρέπει επίσης όμως να κάνουμε είναι δράσεις στον τομέα της δίωξης. Και εδώ να συμφωνήσω με την κυρία Χάνιμπολ, δεν θα φτάσουμε μακριά εάν όχι μόνο δεν ε, διερευνήσουμε ε, την κατάσταση, εάν δεν ψάξουμε, αλλά και αν δεν διώξουμε τους ενόχους. Υπάρχει λοιπόν το σκέλος της διαδικασίας που αφορά την πρόληψη, το οποίο αποτελεί και τη βάση στο κάτω-κάτω της δουλειάς μας, όμως πρέπει να δούμε και τι γίνεται με εκείνους που έχουν κακοποιήσει, έχουν πουλήσει ανθρώπους, γιατί αυτό συμβαίνει. Αγοραπολισίες ανθρώπων. Και πρέπει να παραδεχτώ από τη μία ότι η εμπορία ανθρώπων συνεχίζει να είναι προτεραιότητα, μία από τις πέντε κύριες προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα γίνονται πολλά γι' αυτό, αλλά υπάρχουν και ε, προβλήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, το 7% της χρηματοδότησης πηγαίνει σε δράσεις για την διακίνηση με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό για την διακίνηση παιδιών. Είναι χαμηλότατα τα ποσοστά, ιδιαίτερα για τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εδώ δεν μιλάω μόνο για κορίτσια αλλά και για αγόρια και για άντρες. Όπως σας είπα, το 70% των κονδυλίων προέρχονται ε, από εποχές πριν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν απαγρύπνηση, αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερη δράση. Τώρα, η συνάδελφος από τη Γερμανία έκανε μια ερώτηση και καταρχάς να κάνω μια διακρίνηση. Η Γερμανία μετέφερε ε, όλη την ε, οδηγία το Νοέμβριο πέρυσι, πολύ πρόσφατα. Δεν μπορούσαν λοιπόν να συμπεριληφθούν όλα τα εθνικά μέτρα στην έκθεση. Υπήρχαν μόνο κάποια αρχικά ευρήματα, ε, αλλά δεν είχαμε ακόμα αρκετές πληροφορίες για τη μεταφορά στην νομοθεσία. Όμω τώρα έχουμε αποκρισταλλώσει κάποιε θέσει, έχουμε δει κάποια πράγματα. Καταρχά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση και την εξώθηση στην πορνεία ανθρώπων. Αυτά λοιπόν ε, για την ερώτησή σας. Μετά βέβαια να πω ότι κατέστη επίσης σαφές ότι η πορνεία είναι ένας τομέας υψηλού κινδύνου. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι αρχές επιβολής του νόμου όλων των κρατών μελών, το λέει και η Ευρωπόλ, έχει γίνει η ανάλυση το 2016 σχετική και είναι ε, σαφέστατο το πρόβλημα αυτό. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι όλα τα θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση και τώρα χρησιμοποιώ τα λόγια ενός ανώτατου ε, αξιωματούχου αστυνομικού από την Γερμανία είναι ότι όλα αυτά τα θύματα που εντοπίστηκαν, θύματα εμπορίας ανθρώπων, ε, είχαν διοχετευτεί στην πορνεία. Είναι λοιπόν κάτι που σε καμία περίπτωση δεν είναι αμεληταίο και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη στη δουλειά μας. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η μεταναστευτική κρίση είναι μια τραγωδία. Είναι μια τραγωδία που ε, αφορά όλους, όχι μόνο εκείνους που περνάνε τα σύνορα, αλλά και εκείνους που πέφτουν θύματα εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Σας παρακαλώ όμως να μην ξεχνάτε ότι το δύο, τα δύο τρίτα των θυμάτων είναι Ευρωπαίοι πολίτες που ε, είναι θύματα εκμετάλλευσης εγκληματικών συμμοριών. Να μην ξεχνάμε επίση ότι όσο εμεί τα συζητάμε αυτά υπάρχουν θύματα, είτε πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε όχι, που είναι θύματα. Πρέπει ο νόμος να τους αντιμετωπίζει ίσα και πρέπει να διασφαλίσουμε για αυτούς ε, σαφήνεια, ασφάλεια δικαίου και να υπάρχουν σαφείς ορισμοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Βασιλιάδου. Ευχαριστούμε για την εξαιρετική επισκόπηση και για τις άριστες απαντήσεις που μας δώσατε. Ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχατε. Τώρα να προχωρήσουμε. Σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. τα αποτελέσματα της 61ης ε, συνεδρίασης του UNCSW για την ε, οικονομική ε, ανεξαρτησία και χειραφέτηση των γυναικών. Να καλωσορίσω εδώ τον αναπληρωτή διευθυντή της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ, την υποδιευθυντή, υποδιευθύντρια της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ, την κυρία Χίντι Να της δώσω τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω και εγώ την παρουσίασή μου. Απλώς να παρακαλέσω ποιον ε, είναι υπεύθυνο ε, για τα slides να τα προβάλλει στην οθόνη. Ευχαριστώ και την Επιτροπή που προσεκάλεσε την ε, Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για την ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σας. Όπως ξέρατε, μόλις ήρθα από την σύνοδο που ετησίως λαμβάνει η χώρα στη Νέα Υόρκη και ζητήσατε να σας παρουσιάσουμε τα πορίσματα αυτής της διάσκεψης και στα πλαίσια του High Level Panel επίσης, του πάνελ υψηλού επίπεδου που συνεκάλεσε ο πρώην γραμματέας του, γενικός γραμματέας του ΙΕ για να συζητήσουμε το πώς προχωρούει η επίτευξη των ε, στόχων της χιλιετίας για την ισότητα των φύλων. Λαμβάνοντας υπόψη και τους υπόλοιπους στόχους βάσιμης ανάπτυξης βεβαίως. Αυτό είναι ένα από τα πολλά ε, που, ε, πάνελ που διοργάνωσε η Πατιαρμοστία και επικεντρώνεται στον υγειονομικό τομέα. Γιατί, ε, και υπήρξε μεγάλη εκπροσώπηση στο πάνελ από διάφορου τομεί, με μέλη τη κοινωνία των πολιτών, με συνδικαλιστικέ οργανώσει, με μέλη ε, της ITC, με μέλη από την Ινδία, από πολλές ενώσεις των πολιτών, την Oxfam, τις γυναίκες της απασχόλησης και άλλες οργανώσεις, πολλές κυβερνήσεις και συμπρόεδρος ήταν ο πρόεδρος της Κωνσταντίνα. και ο εκτελεστικός διευθυντής ε, της ε, Λιβετίας ε, από τον επιχειρηματικό κόσμο. Υπήρχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Τανζανίας και άλλες κυβερνήσεις που εκπροσωπούνταν στο πάνελ. Και κάποιες, κάποιοι διεθνείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι προοπτικές ε, και οι οπτικές γωνίες στο πάνελ έρχονταν από τόσο διαφορετικές ε, παρουσίες και πηγές που ήταν πραγματικά φοβερά συνεπαστικό να ακούει κανεί τόση ποικιλία απόψεων αλλά προσπαθήσαμε να πετύχουμε ένα βαθμό συμφωνίας μεταξύ των ε, αποτελεσμάτων στο οποία κατακαλύψαμε. Το μακροσκελές έγγραφο του Σεπτεμβρίου 2016 του ΟΗΕ ήταν βάση των συζητήσεών μας και εντοπίσαμε 7 κινητήριε δυνάμει για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Τα βλέπετε και στο διάγραμμα. Και τέσσερι τομεί όπου πρέπει να εργαστούμε. <clears throat> Τέσσερι τομεί που είναι αλληλένδετοι. Η πραγματική οικονομία, η παράτυπη η παραοικονομία, η γεωργία και άλλοι τομεί έπρεπε να δούμε τι ε, συσχετισμοί υπάρχουν μεταξύ λόγου χάρη νόμιμης οικονομίας και παραοικονομίας ή για την γεωργία και ούτω καθεξής. Η αρχή επί της οποίας συμφωνήσαμε τον πρώτο χρόνο συζητήσεων του πάνελ ήταν ε, ε, ότι το να, μην μείνει κανείς απ' έξω είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να καθοδηγούν τις εργασίες του πάνελ. Δηλαδή, Πρέπει όλες οι γυναίκες να συμμετάσχουν στην ε, επιδίωξη του στόχου SDG 5. Είναι καθοριστική σημασία. Πρόσφατα, τον Μάρτιο, δημοσιεύσαμε την ε, δεύτερη εκθεσή μας για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στον χώρο της εργασίας και που μελετάει τις τέσσερις τομείς εργασίας και τους επτά κινητήρες δυνάμεις που αναφέραμε. Θα έπρεπε να ξεκινήσει στην αρχική σύνοδο, αλλά με τις καιρικέ συνθήκες στην Ευρώπη δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε στη δημοσίευση της έκθεσης. Και τώρα υπάρχει στον ιστότοπο των, ε, ε, του, του, του ΙΕ για τις γυναίκες. Ε, επικεντρωθήκαμε στο μακροοικονομικό περιβάλλον, ένα θέμα που είχε απλώς ε, εξετάσει εκροθυγώς η πρώτη έκθεση, και χρησιμοποιούμε και κάποια από τα συμπεράσματα εργασία εκείνη τη πρώτη συνόδου στην επόμενη έκθεση, την οποία θα αναπτύξω. Ω συνδικαλιστικέ οργανώσει, είχαμε κάποιε πρώτε προτεραιότητε που θα ήθελα να τι αναφέρω και κάποια καλά αποτελέσματα από την 61η Σύνοδο. Πρώτα απ' όλα, το πόσο κεντρική σημασία παίρνει η εξωπρεπή εργασία ε, και η διάσταση τη ισότητα των φύλων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Στα πλαίσια ενό μεταβαλλόμενου κόσμου, χωρίς να δίνουμε έμφαση στην αξιοπρεπή εργασία. Επίσης, θελήσαμε η ποιοτική κρατική εκπαίδευση για γυναίκες και κορίτσια να είναι μια συνιστόσα της όλης προσπάθειας. Είναι σημαντικό από την πλευρά του εργατικού δυναμικού, της ε, εργασιακής δύναμης των γυναικών. Χρειαζόμαστε περισσότερες ε, δεσμεύσεις και αφοσίωση για την κάλυψη του μισθολογικού χάσματος είναι αδιανόητο το 2017 υπάρχει ακόμα αυτό το σοβαρότατο μισθολογικό χάσμα σε όλο τον κόσμο και η κατεύθυνση που βλέπουμε τώρα διαμορφώνεται θα μας πάρει 70 χρόνια για να καλυφθεί αυτό το χάσμα. Και μια από τις βασικές ε, ιδέες είναι ότι η αλλαγή του βιωτικού επίπεδου θα πρέπει να φέρει αλλαγές και στην κοινωνική προστασία και βεβαίως αυτό να ανανεώνει, αλλάζει και τις θέσεις εργασίας που καλύπτουν οι γυναίκες στην ε, αγορά εργασίας. Η εργασιακή διάκριση και ο διαχωρισμό των γυναικών είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συμμετοχή του στην αγορά εργασία. Θέλουμε αναγνώριση των επενδύσεων στην οικονομία των φροντιστών, ώστε οι γυναίκε να είναι ελεύθερε να συμβάλλουν και στις, ε, απασχόληση που παράγει κέρδο και να θεωρούνται παραγωγικέ. Βλέπω εδώ μια βουλευτή με το παιδί της ας πούμε. Το φροντίζει. Είναι μια αναγνώριση του πόσο η δουλειά του φροντιστή που αναλαμβάνουν οι γυναίκε, παράλληλα με όλα τα άλλα που κάνουν, επηρεάζει όλη του τη ζωή. Εδώ θέλουμε και μια αναγνώριση του γεγονότο ότι η βία, ε, η έμφυλη βία, είναι μια από τι πιο σημαντικέ μορφέ βία που δεν λαμβάνεται επαρκώ υπόψη. Και επηρεάζει πάρα πολύ τον χώρο εργασία. Εκεί υπάρχουν και άλλα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί η έμφυλη βία. Και νομίζω ότι ε, έτσι έφτασα στο τέλος των διαφανειών μου. Ε, μου ζητήσατε να παραμείνω σύντομη και θα το κάνω. Ε, μπορούμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ευχαριστώ πολύ. Ήμουν τυχερή και Πήγα και εγώ σε αυτή τη ε, διάσκεψη για λίγες ημέρες. Θα ήθελα να βερθώ στα πορίσματα αυτής της εξποστής πρώτης και συγκεκριμένα σε τρεις πτυχές. Το πρώτο είναι το μισθολογικό χάσμα. Και στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν όμως νομίζω σιγά σιγά αρχίζουμε να επεξεργαζόμαστε έναν ευρύτερο δίκτυο αυτά τις οικονομικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και στον τομέα των συντάξεων. Αυτό αναφέρθηκε στη Νέα Υόρκη. Εκεί περιλαμβάνονται περισσότεροι μισθολογικοί συντελεστές, συνιστώσεις ε, και δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. 39% στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το χάσμα στις συντάξεις. Φανταστείτε τι γίνεται σε λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες. Αυτό λοιπόν το χάσμα ίσως να είναι και χειρότερο. Σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει καν εγγυημένη σύνταξη. Είναι ένας δείκτης που θα ήταν καλύτερος γιατί θα έδειχνε πιο καλά την κατάσταση, αλλά ακριβώς επειδή δεν υπάρχει παντού εγγυημένη σύνταξη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο δείκτης. Το πρόβλημα, όπως είπα, είναι πολύ σοβαρό ιδίω χώρο χώρε που υπάρχει συνταξιοδοτικό σύστημα εγκυμένη σύνταξη, γιατί το μισθολογικό χάσμα είναι μικρότερο από το συνταξιοδοτικό. Και ε, εσεί αναφερθήκατε και σε κάτι άλλο, στου κατώτατου μισθού και την κοινωνική προστασία. Μπορούμε εδώ να καταπολεμήσουμε το μισθολογικό χάσμα με συγκεκριμένα μέτρα. Αλλά σε ό,τι αφορά τη συντάξη, ο βασικό λόγο για την τεράστια αυτή τη διαφορά είναι το γεγονό ότι υπάρχει λιγότερη παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασία, παίρνουν part-time ε, για την ανατροφή των παιδιών του, παίρνουν γονιάδι κτλ. Το κενό αυτό δεν μπορεί να το καλύψουν η τη μυστική κοινωνική προστασία, άρα νομίζω ότι οποιαδήποτε πολιτική κάνει λόγο για συμφιλίωση επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεύτερη πτυχή βία. Μιλήσαμε πολύ για τους ε, ξαναδεστικού γάμους, παιδιών ιδίω, που είναι ένα μείζον πρόβλημα σε πολλές χώρες. Η βία είναι ένα γενικό πρόβλημα βέβαια, το οποίο σοβεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Και νομίζω ότι είναι κρίμα που η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν αναφέρεται στα συμπεράσματα της 61ης αυτής συνάντησης, γιατί είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Ξέρω ότι έτσι γίνεται στο επίπεδο του ΟΗΕ, δεν αναφέρουν δηλαδή άλλες συμβάσεις με το όνομά τους, αλλά θα μπορούσε αυτό το εργαλείο να βοηθήσει να υπάρξουν αλλαγές. Ε, θα έπρεπε νομίζω να αναφέρουμε την Σύμβαση Κωνσταντινούπολη στα συμπεράσματα και που μιλάμε για τη βία. Το τρίτο, εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την ισότητα. Θέλω να αναφέρω μια πτυχή την οποία συζητήσαμε διαμακρών. Το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φίλων τι σημαίνει αυτό. Σήμερα, την ώρα που μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπάρχει πολύ καλή πρόσβαση στην εκπαίδευση για άντρες, γυναίκες και αγόρια, κορίτσια και οι γυναίκες μαθαίνουν πολλά στη ζωή τους, περισσότερα από τους άντρες. Ε, τα στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών όπως είναι το e-banking, το e-shopping, e-selling, e-medicine e-learning. W takich e, obszarach kobiety... Σε όλες αυτές, σε τομείς βλέπουμε ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες αυτές κατά κάποιες ποσοστίες μονάδε λιγότερο συχνά από ότι άντρες. Αλλά με τις τεχνολογίες αυτές πραγματικά θα μπορούσε να γίνει διαφορά και να διευκολύνουμε τη ζωή των γυναικών. Γιατί δεν χρησιμοποιούν λοιπόν οι γυναίκες αυτές τις νέες ευκαιρίες. Κάτι άλλο είναι ότι οι γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες λιγότερο συμμετέχουν από ότι άνδρες στη δημιουργία της ψηφιακής οικονομίας. Πολύ μεγάλο ποσοστό ε, των start-up δεν είναι από γυναίκες. 4% επίσης των ανώτατων κλιμακίων στον τομέα ε, των επιχειρήσεων IT είναι γυναίκες. Σε, αυτά, σε αυτούς τους τομείς λοιπόν βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά ότι ο νέος κόσμος που δημιουργείται, δημιουργείται χωρίς τις γυναίκες. Δεν υπάρχει γυναικεία προοπτική σε αυτόν τον νέο κόσμο. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ψηφιακό χάσμα. μεταξύ των δύο φύλων, που διευρύνεται όλο και περισσότερο όσο περισσότερο αναπτύσσεται ο εν λόγω τομέας, που προσελκύει νέους εργαζόμενους, αλλά αυτοί είναι άνδρες. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και επιτούνται νέα μέτρα πολιτικής. Είναι αυτό νομίζω ένα θέμα που αναγνωρίζεται από πολλούς και θεωρείται πρόκληση για το μέλλον. Και ελπίζω να το αντιλαμβάνεστε κι εσείς και να σας απασχολήσει. Ευχαριστώ. πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ τώρα η Μόνικα Βάνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Διευθύντρια King θα εδώ για να συζητήσουμε την έκβαση της συνάντησης του UNCSW και εγώ στην Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία. Για δεύτερη φορά πηγαίνω στο CSW και ξέρετε ότι για πρώτη φορά είχαμε και ένα ψήφισμα το οποίο είχαμε υπερψηφίσει με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Ήταν μεγάλο, ένα προοδευτικό ψήφισμα και νομίζω ότι σας βοήθησε. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, με εντυπωσίασε Αφενός ε, η ενδυνάμωση, ε, η ενίσχυση ε, που παίρνει κανείς δουλεύοντα με γυναίκες από όλο τον κόσμο για την καθιέρωση διεθνών προτύπων για τα δικαιώματα των γυναικών. Απ' την άλλη, και πάνω σε αυτό θα ήθελα την άποψή σας, ήταν ιδιαίτερο ανησυχητική η κατάσταση που βλέπουμε να πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ήταν σαφές όλες τις συζητήσεις και το είδαμε και στη, σε όλα τα επίπεδα ε, η λογοκρισία ε, και όλα τα άλλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε τα θέματα του οικογενειακού προγραμματισμού, της υγείας, της άμβλωσης κτλ. κτλ. Την έκβαση, την πραγματική έκβαση, πώς την ερμηνεύετε, επειδή έχουμε αυτές τις πολύ δύσκολες νέες συνθήκες. Σημαίνει βελτίωση, πρόοδο αυτή η εξέλιξη. Παραδείγματο χάρη, σε ό,τι αφορά το, τη συμπερίληψη της δέσμευσης του φίλου στην κατάρτιση του προπολογισμού, ε, αλλά έχουμε και άλλα θέματα, πρόσφυγες, SHRH κτλ. Mm. Ε, ε ναι. εντάξει, δεν είναι ημιτοκυβρό στα αγγλικά, δεν μπορώ να κάνω κάποια λαθάκια. Συγχωρέστε με. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την επίθεση που δεχόμαστε, που μας πάει πιο πίσω, πώς μπορούμε να τρέψουμε αυτή την τάση. Γιατί επ' αυτού δεν μπορώ να πω ότι με ικανοποιήσει ιδιαίτερα η έκβαση αυτή της συνάντησης. Με τον Γενικό Γραμματέα είχαμε μια πολύ ε, σημαντική ανταλλαγή απόψεων και η ανάλυση του ήταν άκρος ενδιαφέρουσα. Που είπε δεν έχουμε πρόβλημα τους κανόνες, είτε με τους νόμους, αλλά με την εφαρμογή πιο πολύ. Συμφωνείτε μαζί του, αυτή είναι η ερώτησή μου. Εγώ εν μέρη συμφωνώ για να μην ειλικρινής, γιατί ναι, νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με την εφαρμογή στον ΟΗΕ και όσοι γυναίκε συνεργάζονται, ε, μάλλον εργάζονται στα θέματα διεθνού πολιτική, γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ε, δεν εφαρμόζεται σωστά η πολύ καλή νομοθεσία που έχουμε. Αλλά υπάρχει πρόβλημα έλλειμμα καλή νομοθεσία απ' την άλλη. Και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα επ' αυτού. Um, just wanted to... Κύριε Ward, ε, θέλω να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Στα... Στους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αναφερθήκατε στην χειραφέτηση, στην ανάγκη εκπαίδευση των γυναικών, στο να ενημερωθούν πως πρέπει να προσχωρούν σε συνδικάτα, να οργανώνονται. Ιδιαίτερα σε ορισμένους κλάδους όπου τα δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά όπου οι γυναίκες είναι κακοπληρωμένες, πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Γι' αυτό χαρήκα πάρα πολύ που άκουσα ότι ο συνδικαλισμός είναι καλά οργανωμένος εδώ και χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να προσχωρούν σε συνδικάτα έτσι ώστε να επιμορφώνονται, να ενημερώνονται, διαβίου μάθηση, άτυπη μάθηση. Όλα αυτά είναι θέματα με τα οποία ασχολούνται τα συνδικάτα και οδηγούν στη χειραφέτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Όπως ίσως γνωρίζετε, η αντιπροσωπεία μας συμμετείχε στην 61η Σύνοδο του CHW. Ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν για μας τόσο να επαναλάβουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια θέση που φαίνεται και στο ψήφισμα που εγκρίθηκε το Φεβρουάριο και να εξασφαλίσουμε ότι η θέση αυτή θα διαφαίνεται και στα τελικά συμπεράσματα. Έγινε λοιπόν μια συνάντηση με τις με κυβερνητικές οργανώσεις, με πολλές από αυτές που ήταν παρούσες σε αυτή τη συνάντηση. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι ορισμένες από αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που εκπροσωπούσαν τους πολίτες μας, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πάρα πολύ απογοητευμένες με αυτά τα ε, τα συμπεράσματα. Μας ε, είπαν ότι δεν ελήφθη υπόψη η φωνή των ΜΚΟ. Πώς λοιπόν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αλλάξει αυτή την κατάσταση, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι όταν θα γίνει ετήσια συνάντηση θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην άποψη και τη θέση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και ένα άλλο σχόλιο, επιτρέψτε μου να κάνω, πώς είπε ήδη η συνάδελφος, Συναντηθήκαμε και με τον Γενικό Γραμματέα κύριο Γκουτιέρες, είχαμε μια πάρα πολύ ζεστή συνάντηση, ήταν πολύ ανοιχτή συνάντηση. Και είπε και αυτός με μεγάλη σαφήνεια αυτά που λέμε και εμείς στο Κοινοβούλιο. Βλέπουμε δυστυχώς όμως μία υπαναχώρηση, ένα πισωγύρισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Δεν πάμε μπροστά. Και μάλιστα γνωρίζουμε και όλες ότι ορισμένα κράτη-μέλη έλαβαν τέτοιες αποφάσεις που είναι ξεκάθαρο ότι κάνουν βήματα προς τα πίσω. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε δεδομένων όλων αυτών. Πώς μπορούμε τουλάχιστον να διατηρήσουμε το status quo. Σήμερα εγκρίθηκε και το κείμενο μιας προφορικής ερώτησης προς το Συμβούλιο και σε αυτήν την ερώτηση ζητάμε να μάθουμε πώς ερμηνεύει το Συμβούλιο αυτές ε, τις, ε, αυτά τα συμπεράσματα και αν η θέση μας ε, διαφαίνεται σε αυτά τα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν εξαιρετικές οι ερωτήσεις σας. Θα αρχίσω λοιπόν με την ερώτηση για τα αποτελέσματα και θα το πάρουμε από εκεί. Και θα ήθελα να πω ότι όταν ε, φτιάχναμε αυτές τις διαφάνειες ακόμα ήταν υποδιαπραγμάτευση τα σημερινά του Συμβουλίου, δεν τα γνωρίζαμε. Και μάλιστα όταν φτιάχνουμε τις διαφάνειες της παρουσίασης νομίζαμε πως δεν θα υπάρχουν καν συμπεράσματα. Ήταν, πότε ήταν, Παρασκευή, πρωί, Παρασκευή, απόγευμα. Ακόμα είχαμε 30 παραγράφους υποδιαπραγμάτευσης και ο Πρόεδρος ήταν έτοιμος να παρουσιάσει μία δήλωση χωρίς αυτές. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, ε, αυτό που σημείωσα εγώ ήταν ε, ότι το κείμενο των συμπερασμάτων είναι καλό, πολύ καλό μάλιστα σε ορισμένα σημεία, εξαιρετικά προβληματικό σε άλλα και ε, δυστυχώς δεν καταφέρνει να ε, κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Όντω υπάρχει οπισθοχωρήση σε ορισμένα κράτη-μέλη, όντω υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Ε, τώρα, μα είπατε, ίση αμοιβή για ίση εργασία. Συμφωνώ μαζί σα απόλυτα. Αυτό το συζητήσαμε και όταν κάνουμε λόγο για το μισθολογικό κενό πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκε ε, που παίρνουν σύνταξη, σταματούν την εργασία τους εξαιτία αυτού του μισθολογικού κενού. Πολλές φορές, ε, μάλιστα, πολλές γυναίκες σταματούν να εργάζονται για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, για να φροντίσουν μέλη της οικογένειας, για να αποφύγουν την επισφαλή εργασία κτλ. Όμως αυτή η απλή φράση, ίση δουλειά για ίση εργασία, μην νομίζετε πως ήταν τόσο εύκολο να συμπεριληφθεί. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, α πούμε, δεν, έχουν αυτό, δεν ακολουθούν αυτό το σκεπτικό. Μιλάνε μόνο για ίση αμοιβή, όχι για εργασία ίση αξία, Δεν, δεν αναφέρονται σε ίση αξία. Αυτό λοιπόν ε, δεν είναι θέση των ΗΠΑ, δεν είναι θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν είναι μάλιστα θέση πολλών κυβερνήσεων. Το πώς δηλαδή υπολογίζεται η αξία της εργασίας των γυναικών έτσι ώστε να κλείσει αυτό το μισθολογικό χάσμα. Τώρα ε, αναφερθήκαμε στους ε, κατώτατους ε, βασικούς μισθούς που είναι αξιοπρεπείς, που σου επιτρέπουν να ζήσεις. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και στις συντάξεις, να, αναφερθούμε στο πρόβλημα, στο χάσμα που υπάρχει στις συντάξεις. Πρέπει να δούμε όλες τις πτυχές του γιατί οι γυναίκες είναι εκτός αγοράς εργασίας για παράδειγμα, θα μπορούσαν οι γυναίκε όσο δεν εργάζονται για να φροντίσουν διάφορα μέλη τη οικογένεια, να, έχουν ασφαλιστικές εισφορές για τη σύνταξη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό να κοιτάξουμε επίσης και τι διαφορέ από χώρα σε χώρα και από περιφέρεια σε περιφέρεια. Χρειάζεται να τεθούν επίσης κάποια ανώτατα όρια που θα ισχύουν καθολικά ένα βασικό ε, κατώτατο επίσης όριο κοινωνικής προστασίας για να αντιμετωπιστούν αυτά τα μισθολογικά χάσματα. Μετά, υπάρχουν σίγουρα αρκετοί νόμοι με προβληματική εφαρμογή που επιβραδύνει την πρόοδο. Τώρα υπάρχει πρόοδος, εγώ θα έλεγα όχι. Εδώ δεν υπάρχουν αρκετές πολιτικές, ε, μακροοικονομικές πολιτικές για παράδειγμα αυτός ο τομέας ε, είναι ένας προβληματικός τομέας με την έννοια ότι οι κυβερνήσεις ε, εθελοτυφλούν σε θέματα ισότητας και όταν καταρτίζεται μια μακροοικονομική πολιτική η οποία συνεισφέρει στο ΑΕΠ, ή μάλλον η εργασία των γυναικών συνεισφέρει στον ΑΕΠ, αλλά δεν συνυπολογίζεται σε αυτή τη μακροοικονομική πολιτική. Εάν υπήρχε μια μακροοικονομική πολιτική που θα λάμβανε υπόψη τα ζητήματα ισότητας, για παράδειγμα ε, η δουλειά που κάνουν οι γυναίκες πέρα από την εργασία, στο σπίτι, στη φροντίδα άλλων. Είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να συνεκτιμηθεί έτσι ώστε να κλείσει αυτό το κενό. Μετά, οργάνωση. Σίγουρα και εγώ από συνδικάτο προέρχομαι, οπότε αναγνωρίζω απόλυτα το πόσο σημαντική είναι η οργάνωση. Χρειάζεται λοιπόν δουλειά με τα συνδικάτα να ενισχυθεί το δικαίωμα του να συμμετέχει σε συνδικάτο, να κλείσουν όλα αυτά τα κενά, το μισθολογικό κενό ας πούμε. Χρειάζονται συλλογικές διαπραγματεύσεις, συνδικαλισμός των γυναικών με αυξημένα ποσοστά συνδικαλισμού στις γυναίκες θα μειωθούν σίγουρα ε, τα, οι μισθολογικές ανισότητες. Υπάρχουν όμως και εδώ προβλήματα, μην νομίζετε, που μας κρατάνε πίσω. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω ε, για να αλλά να σταθώ σε τρία πράγματα. Στον ε, ρόλο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, καταρχάς. Να πω ότι η συνεργασία ήταν εξαιρετική ε, ανάμεσα στα Ηνωμένα Έθνη και στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Ε, αναγνωρίστηκε η ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού και πιστεύω πως η συνεργασία μας με τη Διεθνή Οργανώση Εργασίας αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα του πόσο καλά μπορούμε να δουλέψουμε. Ε, βέβαια, πολλές κυβερνήσεις ε, είπαν γιατί τη δουλειά έχουν αυτοί εδώ. Όμως ε, φυσικά και έχουν στην παρακολούθηση της εφαρμογής τον έλεγχο και θα συνεχίσουμε λοιπόν την καλή συνεργασία με αυτούς. Μετά, η γεωπολιτική ήταν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων να πω. Δεν θέλω να δείξω με το δάχτυλο αντιπροσωπείες και να αναφερθώ με ονόματα, αλλά υπήρχαν ορισμένοι που υιοθέτησαν πολύ επιθετική στάση. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ την ε, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν, οι οποίοι ήταν υποστηρικτικοί τόσο σε εμά ως συνδικάτα όσο και γενικότερα στο, στα αιτήματα αυτά για ισότητα. Ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό για τη δουλειά μας να φτάσουμε σε ένα στάδιο που θα έχουμε μεγάλους οργανισμούς όπως εσείς που θα μας βοηθούν στην άσκηση πίεσης. Επίσης, ε, πρέπει να μιλήσουμε για πολλά ακόμα, να μιλήσουμε για τις ε, αξίες της οικογένειας, να υπάρχει διαμεσολάβηση, να τονιστεί η σημασία ε, αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα περιοριστώ εδώ για να μην καταναλώσω άλλο χρόνο και θα σας ευχαριστήσω όλη μία φορά για την πρόσκληση. Ευχαριστώ να συνεχίσουμε. Έχουμε δύο ακόμη σημεία στην εμείς διάταξη. Το σημείο 8. Έκθεση για την αποστολή στη Μάλτα 2017. Θα βρείτε το τι έγινε στη Μάλτα στα έγγραφά σας 2 με 4 Φεβρουαρίου. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, θεωρείται εγκεκριμένη η αναφορά αυτή. Και μετά έχουμε το επόμενο σημείο τα σοφρονιστικά ιδρύματα και οι συνθήκε που κρατούν εκεί. Σχέδιο γνωμοδότηση από την κυρία Ματέρα, η οποία δεν μπορεί να παραστεί σήμερα. Και κανείς δεν είναι εδώ για να την αντικαταστήσει. Οπότε δεν θα εξετάσουμε την έκθεση τώρα. Μπορείτε να τη διαβάσετε αν θέλετε. Και να πω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 31 Μαρτίου το μεσημέρι. Στις 11 Μαΐου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα ψηφίσει στις 29 Μαΐου. Και το έγγραφο θα περάσει από την Ολομέλεια τον Ιούλιο του 2017. Να ευχαριστήσω όλους και όλες και να θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 11 και 12 Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ και την γραμματεία. Ευχαριστώ. Yeah, yeah. Ah, ah, a little later, yeah. <laughs> okay.